ΕΝΕΦ έλαβα αιτήματα διορισμού και αλλαγών στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες. Όλα αυτά θα μπουν στα πρακτικά της σημερινής ε, συνεδρίασης και εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της έγκρισης των πρακτικών θεωρούμε πως εγκρίνονται αυτοί οι διορισμοί και οι αλλαγές. Επίσης, να ενημερώσω το σώμα πως ε, μαζί με